So, hello everybody. It's a pleasure. Καλησπέρα σας και με χαρά σας καλωσορίζω εδώ. Uh, as this meeting is web streamed, hopefully. Uh, it's a pleasure for me. Με χαρά λοιπόν σας καλωσορίζω στη δημόσια ακρόασή μας για τα... για τα κρατικά είχε συμφωνηθεί πέρυσι να γίνει με τέτοια ακρόαση, μια και ε, ενδιέφερε όλους μας. Χαίρομαι λοιπόν που κηρύσσω την έναρξη τη ε, ακρόαση Το θέμα των κρατικών κρατικών επενδύσεων έχει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τη σημασία και το ρόλο που αυξάνονται εκθετικά των, ε, των επενδύσεων αυτών. Μιλάμε για 5 έως 8-3 ε, δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδα ανάλογα και με τον ορισμό που επιλέγουμε. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροοικονομική διαχείριση και στην α, οικονομική σταθερότητα και συνδέεται αυτό με τα δημοσιονομικά, με τους κανόνες ε, που τους διέπουν σε ό,τι αφορά τους ε, κανόνες και τις συνθήκες ρευστότητας, καθώς και με τις αποκλήσεις σε ό,τι αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο η πολιτική λοιπόν σε ό,τι αφορά τις κρατικές αυτές ε, ε, επενδύσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτές τις ε, διαστάσεις. Και επίσης η κρατική πολιτική θα πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες της και να την ε, διανέμει σωστά μεταξύ των διάφορων δοσμικών οργάνων, να διαφαλίζει δε και την ανεξαρτησία των οργάνων αυτών. Και ο στόχος λοιπόν της συνεδρίασης της ΕΚΟΝ σε ό,τι αφορά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα στρατηγικά επενδυτικά ταμεία είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον λειτουργούν σωστά, με σωστή διαφάνεια και κατά πόσον κατανοούμε τις συστημικές επιπτώσεις ε, για τις αγορές των κρατών που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Και ο παράγοντας ε, σταθεροποίησης, ο παράγοντας της αυξημένης α, ε, μεταβλητότητας. Καθώς και την, το ρόλο των ε, κυβερνήσεων ως ε, φορείς που συμμετέχουν στην αγορά. Επίσης, στρατηγικά επενδυτικά ταμεία και οι επενδύσεις αυτές κατά πόσο θα μπορούσαν να συνδράμουν μακροπρόθεσμα σε πιο πολλές επενδύσεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις επενδύσεις. Πρωτού δώσουμε λοιπόν το λόγο στους πανελίστες μα να σα παρουσιάσω ποιοι είναι. Με χαρά καλωσορίζω τον κύριο Τόρε Φαμπράκ, ο οποίο είναι ήδη υπουργό στο ε, Υπουργείο Οικονομικών στην Νορβηγία το 2015. Το, ταμείο, το Υπουργείο Οικονομικό α, επιβλέπει το συνταξιδοτικό ταμείο τη Νορβηγία, το οποίο είναι το πιο μεγάλο στην Ευρώπη, 900 δι ε, δολάρια στις αρχές του 2017 ελπίζω να στέκουν τα στοιχεία αυτά. Ελπίζω να καλωσορίσω και τον κύριο Γκουίντο Πικισάο. Ναι, σας ζητώ συγγνώμη για την τραγική προφορά μου. Ε, είναι διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο τμήμα θεσμικών, θεσμικής στρατηγικής που είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τα στρατηγικά επενδυτικά ταμεία. Και με μεγάλη μου χαρά επίσης καλώ ορίζω και πάλι στην Επιτροπή μας την καθηγήτρια Στέφανη Γκρίφιθ Τζόνς, η οποία έχει έρθει και άλλες φορές στην Επιτροπή μας, γνωστή ακαδημαϊκή, για θέματα μακροοικονομικής. Είναι διευθύντρια των προγραμμάτων οικονομικών αγορών στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και έχει κάνει διάφορες και πολύ άριθμες δημοσιεύσεις για τα θέματα αυτά. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους σας από πλευρά μου. Έχουμε Δυστυχώ αυτηρού κανόνες σε ό,τι αφορά το χρόνο ομιλία, ε, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Να σας δώσω 10 λεπτά για τα εισαγωγικά σας σχόλια και μετά θα έχουμε το γύρο των έρωτα απαντήσεων με τα μέλη της Επιτροπής μας, τους Ευρωβουλευτές. Όπως σας ε, αν συμφωνείτε, θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που αναφέρεστε και στο πρόγραμμα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον πρώτο μας πανελίστα. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω στο πάνελ αυτό. Πρόκειται για μέσα ειδικού σκοπού, πολλοί έτσι τα ορίζουν, το οποίο διαχειρίζονται εθνικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν ε, από 80 τέτοια ταμεία, τα οποία είναι 10% της συνολικής αγοράς εισαγμένων equities και ομολόγων. Πάνω από, από το μισό του κεφαλαίου βασίζεται σε τέτοια funds. Τα μεγαλύτερα τέτοια funds βρίσκονται στην Νορβηγία, την Κίνα, το Μπουντάμπι, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τη Σιγκαπούρη και το Κατάρ χώρες που είναι ετερογενείς ε, όσον αφορά και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν εξελιχθεί και το πολιτικό επίσης πλαίσιο, αλλά έχουν και διαφορετικές ε, διευθετήσεις όσον αφορά την διαφάνεια. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το ζήτημα και να τα δει σαν ένα σύνολο επενδυτών. Γι' αυτό και εγώ θα περιοριστώ σε ζητήματα κλειδί που έχουν να κάνουν με την ε, Νορβηγία και το δικό μας τέτοιο παιδιτικό ταμείο που ονομάζεται Government Pension Fund Global. Αρχίσαμε από το 2008 με 24 αρχές και πρακτικές όσον αφορά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία που είναι διαφάνεια, η καλή ε, διακυβέρνηση, η λογοδοσία και συνετές επενδυτικές πρακτικές. Και παρόλο που συμμετέχει στο Διεθνές φόρου Επενδυτικών Κρατικών Ταμείων η Νορβηγία, εμείς στηρίζουμε το έργο του φόρουμ αυτού για την προώθηση και των αρχών του Σαντιάγο, που αποτελούν ελάχιστες προδιαγραφές. Στη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη έχει μεγάλο ρόλο η διαφάνεια και ο στόχος των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολιτικές από μια μεριά ε, φιλοδοξίες και από την άλλη μεριά υπάρχει και ο χρηματοπιστωτικός στόχος. Το ταμείο μας λοιπόν αρχικά ονομάστηκε Norwegian Petroleum Fund επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το φυσικό πόρο και το χρησιμοποίησαμε σαν ένα μέσο για να ξεχωρίσουμε τα μεταβλητά έσοδα από τις τρέχουσες ε, δαπάνες και δημιουργήθηκε το 1990 το ταμείο αυτό. Δύο δεκαετίες δηλαδή αφού του ξεκίνησε η παραγωγή πετρελαίου. Και τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στο ταμείο και κάθε χρόνο μεταφέρονται στο προπολογισμό μας. Ε, μεταφέρεται και επενδύεται κεφάλαιο από το ταμείο αυτό στο εξωτερικό. Με, έχοντας υπόψη μας και πολιτικές παραμέτρους, αλλά βέβαια και χρηματοπιστωτικές. Θέλουμε να είμαστε ένας μεγάλος διεθνής επενδυτής. Τώρα θα σας μιλήσω για την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου μας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένας βαθμός κινδύνου και πρέπει να τον αναλάβουμε αυτό. Και γι' αυτό υπάρχει κάθε φορά το λεγόμενο risk profile. Είναι απαραίτητο αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Ταμείο πάντα στην ίδια πορεία. Ε, για μας ο βασικός εταίρος είναι το Νορβηγικό Κοινοβούλιο και βέβαια και οι πολίτες της Νορβηγίας, στους οποίους ανήκει το επενδυτικό αυτό ταμείο τελικά. Ο Υπουργό Οικονομικών έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του ταμείου αυτού, αλλά λειτουργικά τη διαχείριση την έχει αναλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα, η Norges Bank. Το Υπουργείο θέτει κάποια κριτήρια λοιπόν για αποκλήσεις από τον δίχτυ όσον αφορά το ταμείο μας. Έτσι υπάρχουν περιορισμοί και σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς λαμβάνονται στο Υπουργείο διαχειριστικές αποφάσεις. Βέβαια, οι επενδύσεις στις διάφορες χώρες δεν είναι ανεξάρτητες από τις πολιτικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν απόδοση με ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο θεωρείται αποδεκτό από τους ιδιοκτήτες. Το Ταμείο λοιπόν τυχαίνει χρηστής διαχείρισης και υπεύθυνη. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν την ανάμιξη της πολιτικής, αλλά ότι πρόκειται για μια προϋπόθεση προκειμένου να ακολουθεί τους κανόνες που έχουν τεθεί το Ταμείο και να θεωρείται νόμιμο. Το επίπεδο κινδύνου πρέπει να είναι αποδεκτό από τους Νορβηγούς. Το Ταμείο, πρέπει να σας πω, ότι δεν ακολουθεί περιβαλλοντική πολιτική, ούτε είναι μέσο εξωτερικής πολιτικής. Οι επενδύσεις μας είναι είτε εισαγμένο στο χρηματιστήριο έκοτης είτε άλλα μέσα, ε, υποθήκες, φροντίζοντας να υπάρχει μια, ένας, ε, σε επέκταση που να καλύπτει πολλές γεωγραφικές περιοχές, χώρες, κλάδους, εταιρείε, προκειμένου ακριβώ να μειωθεί ο κίνδυνος. Αποτελεί λοιπόν έναν επενδυτή το ταμείο μας, σε σχέση με 9.000 περίπου εταιρείε και 1.200 εκδότες τίτλων. Επίσης, η στρατηγική μας ε, βρίσκεται σε 62,5% του benchmark index που λαμβάνει υπόψη της equities. Και αν συγκρίνουμε με το χαρτοφυλάκιο το συνολικό, το ταμείο μας εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγμένες equities και λιγότερο σε επενδύσεις ομολόγων βάσει του επενδυτικού μας ορίζοντα και κάθε φορά εξισορροπούμε τα πράγματα για να μην αποκλίνουμε πάνω από 4% από τον αρχικό μας στόχο. Όταν βέβαια πέφτουν οι μετοχές στο ταμείο μας, φροντίζει να προσφέρει ρευστότητα, αγοράζοντας εισαγμένες equities. Και παίρνουμε και ομόλογα για παράδειγμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια πολιτικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ώστε να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Έτσι θα διασφαλίσουμε την αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου κινδύνου, κάτι το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν πάντα οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Εσημορφόμαστε με τις απαιτήσει του Σαντιάγο για τη διαφάνεια και η επενδυτική εντολή του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι πρέπει να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα στα όρια που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. Όλοι όσοι έχουν τίτλους πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως. Η διαφάνεια επίσης σημαίνει να καταλάβουμε και πώς γίνεται η διαχείριση του ταμείου αυτού. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφάνεια όσον αφορά τις επενδύσεις μας, όλα τα έγγραφα, όλες οι αναφορές δημοσιεύονται στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Νορβηγικής Τράπεζας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σεβαστήκατε απολύτως το όριο του χρόνου που σας διέθεσα. Δεύτερος ομιλητής τώρα στο πάνελ είναι ο Γκουίντο Μπικιζάου. Παρακαλώ, Γκουίντο. Ευχαριστώ, κύριε Φέρμπερ, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τιμή μου που έχω προσκληθεί να μιλήσω για τα ταμεία του κρατικού πλούτου. αυτή η κατηγορία επενδυτών χειρίζονται περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 7-3 δολάρια και είναι προφανής η μεγάλη σημασία τους. Στι σύντομε παρατηρήσει μου θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερι βασικού τομεί που από την εμπειρία μα ξέρουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη για να καταλάβουμε τη σημασία και το περίπλοκο των SWF Συγκεκριμένα την διάθεση για επενδύσεις και την αντίκτυπο στην αγορά, την τεχνογνωσία και την δέος επιμέλεια, την διακυβέρνηση και τη σύγκρουση συμφερόντων και τα κονδύλια, τα ταμεία αυτά ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πρώτα απ' όλα η διάθεση για επενδύσεις και ο αντίκτυπος στην αγορά. Αυτά τα κονδύλια θεωρούνται μακροπρόθεσμοι επενδυτές και επιτρέπουν περισσότερο από τους μέσους επενδυτές μεγαλύτερο κινδύνου επενδύσεις χαρακτηρίζονται από μια αργή διαδικασία ε, και έχουν ένα μακροπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Το ίδιο και η μεταβλητότητα της αγοράς και πώλησης των διαδικασιών των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των SWF αυτό, καθώς οι σχετικές στατικικές ε, καθοδηγούνται όχι από τις ε, βραχυπρόθεσμες επιστροφές, αλλά γι' αυτό δεν επηρεάζονται και τόσο πολύ από τις βραχυπρόθεσμες δικημάνησες στις τιμές. Η ίδια η φύση των ε, ταμείων αυτών δεν οδηγεί σε απεπένδυση ε, μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες και αυτό ε, όταν υπάρχει μια σχετική στατηγική εμπορίας. Αυτό εξηγεί γιατί οι σχετικές επενδύσεις γίνονται κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία ακίνητα και σε υποδομές. Επίσης μπορούν να διαιρεθούν σε εμπορικά και μη εμπορικά κονδύλια οι επενδύσεις αυτές κατά ε, πλειοψηφία παρουσιάζουν τη δυνατότητα απεπένδυση για να σταθεροποιηθούν οι διακυμάνσει των τιμών. Το δεύτερο στοιχείο είναι η τεχνογνωσία και η δέουσα επιμέλεια. Ε, η ρεσιμότητα για τις επενδύσεις όταν ε, παραχωρείται η δυνατότητα επένδυσης έχει να κάνει με τις κρατικές προτεραιότητες και δεν είναι απλώς οικονομικοί οι όροι που λαμβάνονται υπόψη. Με συγχωρείτε. Με Εάν λοιπόν τα SWF είναι μακροπρόθεσμα σταθερή επενδυτική μορφή, η δυνατότητα να αποφασίσει κανείς σαφής ε, σαφείς στρατηγικές επένδυσεις είναι στον πυρήνα των ερωτήσεων για το κατά πόσο μπορεί να προκληθούν ε, συστημικοί κίνδυνοι. Η εμπειρία μας δείχνει ότι κάποια από αυτά τα κονδύλια, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και την τεχνογνωσία της επένδυσης δεν έχουμε ακόμα προηγμένη γνώση. Από έναν αριθμό SWF βλέπουμε ότι οι αποφάσεις για επενδύσεις ακολουθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι εις βάθος ανάλυση των σε στοιχείων όπω ορίζονται για τι επενδύσει. Σε κάποιε περιπτώσει τα SWF ε, εκχωρούνται σε ένα τρίτο μέρο για να προκαλέσει ή να, ε, πυροδοτεί, να ενεργοποιήσει τι επενδύσει βάσει προσυμπεφωνημένων αρχών ε, με την αρχή τη δεούσα επιμέλεια. Ω προ τη διακυβέρνηση και τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο χώρο στον οποίο χρειάζεται περισσότερη πρόοδο είναι η διακυβέρνηση και η διαφάνεια. Το 2008, 30 από αυτά τα φαντ που συνολικά εκπροσωπούν το 80% των περιουσιακών ε, στοιχείων που ε, διαχειριζόμαστε ε, έπρεπε να υποβληθούν στι αρχέ τη διαφάνεια, τη κυβέρνηση λογοδοσία και των προληπτικών επενδυτικών πρακτικών, τη λεγόμενε αρχέ του Σαντιάγκο. Η ομάδα εργασία που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό μεταβλήθηκε στο, στο Διεθνέ Φόρουμ των SWF, που προωθεί την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο για τι κοινέ αρχέ και διευκολύνει την κατανόηση των SWF και των δραστηριοτήτων του βάσει των αρχών του Σαντιάγκο. Παρά την προσχώρηση σε αυτέ τι αρχέ, παρόλα αυτά, η εμπειρία μα δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλε ανισότητε μεταξύ των διάφορων funds, στον τρόπο δηλαδή που υλοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές και διασφαλίζεται η διαφάνεια. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ακόμη ε, διαπλοκή μεταξύ των αποφάσεων για επενδύσεις και των κρατικών συμφερόντων. Οι πολιτικοί στόχοι που αναμένεται να εκπληρώσουν τα SWF δεν είναι σαφώς τεκμηριωμένοι και αυτό ε, ε, εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα κάποιων επενδύσεων και για κάποιες πολιτικές απεπένδυσης. Η αιρεσιμότητα των επενδύσεων όταν η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων εκχωρείται σε τρίτους περιλαμβάνει όρους που έχουν να κάνουν με στόχου ε, κρατικού χαρακτήρα και όχι μόνο με οικονομικά συμφέροντα. Αυτό μπορεί λόγω χάρη να έχει να κάνει με τι διασυνδέσει μεταξύ εθνικών εταιριών, κρατικών δηλαδή εταιριών και περιουσιακών στοιχείων, η έλλειψη διαφάνεια και σαφών πολιτικών στόχων έχει μεγάλη επιρροή στη διακυβέρνηση των ταμείων αυτών και στο πώς γίνονται αντιληπτά ω προ τα πρότυπα που εφαρμόζονται. Ε, εδώ ο μοναδικό χαρακτήρα των SWF πρέπει να συνδυαστεί με, το, με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και κοινού πολιτικού στόχου. Εάν δεν υπάρχει αυστηρή διαχείριση κάποιων από τα SWF, δεν θα υπάρχει και απόλυτη ανεξαρτησία από τι δικέ του τι κυβερνήσει, ε, ώστε αυτό θα ρίξει σκιέ στην ενδεχόμενη χρήση για, μεγαλύτερες, ε, για μεγαλύτερα επιτεύγματα και λόγω τη ιδιαίτερη επενδυτική φύση αυτών των ταμείων. Τέλος, για τα SWF όταν είναι εταίροι και συμμετέχουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Από όσα είπα, η ίδια η φύση των SWF είναι μεικτή, είναι δυτή. Δηλαδή συμπεριλαμβάνουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Πρώτον, μια σαφή μακροπρόθεσμη ε, λειτουργία, δηλαδή δυνατότητα απορρόφησης ε, περιορίζοντας την ε, επένδυση σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία και μετά μια σχετικά όχι δυνατή διακυβέρνηση που περιορίζεται λόγω τη δέσμευσης επιμέλειας και τη σχετική τεχνογνωσία. Ενώ το πρώτο χαρακτηριστικό κάνει τα SWF ιδανικά ως συμμετοχή σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το δεύτερο εγείρει ερωτήματα για το ποια ποιε διαδικασίε πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σχετιστούν με στρατηγικέ επενδύσει. Σε ορισμένε περιπτώσει, τα SWF έχουν ε, ε, συμπεριληφθεί σε ε, συμφωνίε για να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμε επενδύσει με πολυμερεί τράπεζε. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει, λοιπόν, υπάρχουν συμφωνίε και ε, προσυπογράφουν ένα μέρο των περιουσιακών του στοιχείων που έχει ξεκινήσει από μια πολυμερή τράπεζα βάσει συγκεκριμένων προποθέσεων τη στιγμή της σύναψη της συμφωνία. Η πολυμερή διάσταση ε, είναι που η τράπεζα είναι αυτή που τηρεί τα αρχεία και διατηρεί πλήρη ευθύνη για τις πιστώσεις που έχουν ε, σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία γίνεται η επένδυση. Η έμεση ε, προσδοκία είναι ότι η πολυμερής τράπεζα με την τήρηση αρχείων θα πετύχει να διαπραγματευτεί κατάλληλους όρους σε περίπτωση γεγονότων πιστοτικών και θα μειώσει στο ελάχιστο κάθε δυνατότητα απολειών που έχουν να κάνουν με το Ταμείο, ακριβώς λόγω της μοναδικής της πιστοδοτικής ε, δυνατότητας. Αυτές οι προσδοκίες δημιουργούν τις εξής, ε, τις εξής ε, συνέπειες κινδύνους όπως τη λογοδοσία και την θύμη των SWF. Δηλαδή η απόφαση να διαπραγματευτεί κανείς τους όρους μπορεί να μην είναι η καλύτερη από οικονομικής άποψης και να λαμβάνονται υπόψη και άλλες μέρημνες όπως κοινωνικές ή περιβαλλοντικές. Επιπλέον δεν είναι σαφές αν οι προϋποθέσεις που από τα α, ε, ταμεία αυτά για να ε, αποδώσουν πόρους ε, σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ξεκινήσει από πολυμερείς πηγέ, πηγές διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του στη δέωση επιμέλεια και την διαδικασία επιλογής. η διαδικασία επιλογής πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένη απόφαση από το φαντ να δεχτεί μια ε, επένδυση. Αλλά εμέσω μπορεί να επηρεάζεται από την πολυμερή ε, τράπεζα και να μην είναι ανεξάρτητη η επιλογή των ε, προγραμμάτων που θα επιλεγεί να χρηματοδοτηθούν. Αυτό δημιουργεί κινδύνους ως προς την φήμη των SWF. Επίση, η προτιμησιακή δυνατότητα διατυπωμάτευση ευνοϊκότερων όρων είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη και μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίε ιστορικά. Οι πολυμερεί τράπεζε έχουν διασφαλίσει επικοδομητικό διάλογο με κυβερνήσει και αρχέ σε περίπτωση πιστοτικών γεγονότων για περιουσιακά στοιχεία που έχουν σοβαρό αντίκτυπο, εμέσω ή αμέσω, στην ε, δημόσια διοίκηση μια χώρα. Τόσο διάλογο ε, υπονοεί ότι οι πολυμερεί τράπεζε έχουν μια αποτιμησιακή σχέση, η οποία θεωρείται αποδεκτή και επιθυμητή. Επειδή οι πολυμερεί τράπεζε έχουν ε, οριοθετημένο ισολογισμό και μπορούν τα και μπορούν συγκεκριμένα περιουσιακά του στοιχεία να τα χειριστούν προτιμησιακά. Όμω οι πολυμερεί αναμένεται να στηρίξουν και του ε, δανειζόμενου σε δύσκολε συνθήκε ε, και να συνεργάζονται στενά με τι κυβερνήσει σε περίπτωση που ε, διαταραχθούν οι οικονομικοί όροι μια επένδυση. Αυτή η εταιρική σχέση ή η συμφωνία εκχώρηση που θα ήταν υποφελή για τα SWF λόγω τη ιδιαίτερη φύση των πολυμερών δραστηριοτήτων του έχουν να κάνουν και με το συνολικό μέγεθο των περιουσιακών στοιχείων και από το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια διαδικασία να καμψήσει ένα επαρκή διάλογο ανάπτυξη. Να ολοκληρώσω. Ε, βλέπουμε ότι πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένε πρακτικέ για την εταιρική σχέση επενδύσεων με τα SWF, διασφαλίζοντα πλήρη ανεξαρτησία στον κύκλο δημιουργία και ε, αλληλοσυσχέτιση των μακροπρόθεσμων εταίρων, από οι πολυμερεί τράπεζε. Αυτή η ανεξαρτησία θα επιτρέψει να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι όπω έχουν οριστεί από τι κυβερνούσε αρχέ. Επιπλέον, θα πρέπει η ανεξαρτησία να είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για να μην υπάρξει κίνδυνο προ τη φήμη των SWF δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για να ληφθούν σωστέ πολυμερεί αποφάσει. Αυτό πρέπει να ισχύει ιδίω στην περίπτωση που ε, οι πόροι των SWF κατευθυνθούν στο ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων ε, του Γιούνκερ, του οποίου ανεξαρτησία ε, με συγκεκριμένε πρακτικέ πρέπει να προστατευτεί. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει διαρκή διάλογο με τα SWF και όλο ιδιαίτερο με αυτά που έχουν αποδείξει ότι έχουν καλύτερη διακυβέρνηση και περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό θα είναι πολύτιμο ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε τι κατάλληλε πρακτικέ για να συσχετίσουμε τι μακροπρόθεσμε επενδύσει των SWF μαζί με του μακροπρόθεσμου οικονομικού στόχου και πρωτοβουλίε που έχουμε, όπω το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τελευταίο. Τελευταία μάλλον. Η Stephanie Griffith Jones που μελετά ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η εξέλιξη των ε, ταμείων ε, κρατικών, κρατικού, ε, κρατικών ταμείων και οι σχετικές εφαρμογές τους και κάποιες εφαρμογές στην ε, στρατηγικές ε, επενδύσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, σας έχω στείλει και κάποια, κάποιους πίνακες, κάποια γραφήματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι αρχικά τα ταμεία αυτά αναπτύχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ήταν υψηλές ε, οι τιμές των πρώτων υλών και Το 2007, για παράδειγμα, είχαν φτάσει σε επίπεδο περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 10 χρόνια αργότερα είχαν φτάσει τα 7,5-3 δολάρια. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ωστόσο, και αυτό που φαίνεται και στον πίνακα, στο γράφημα, είναι ότι καθώ οι τιμές από τον πρώτο υλών έπεσαν δραστικά το 2010, και πολλές ε, από τις χώρες είχαν μεγάλα ε, πλεονέσματα τρέχοντων λογαριασμών τα οποία συρρυκνώθηκαν. Οι πόροι αυτοί δεν ε, περιορίστηκαν αντίστοιχα, όπως βλέπετε παρακάτω στον πίνακα. Από το 2014 μέχρι το 2016 ήταν μικρή η μεταβλητότητα σε ό,τι αφορά το συνολικό όγκο των ταμείων αυτών. Αυτό φαίνεται και στον πίνακα και στο γράφημα. Και θα επανέλθω σε αυτή την ανησυχία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις πωλήσει αυτών των ε, ταμείων ε, που πιστεύω ότι είναι υπερβολικές. Να πω επίσης ότι παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι τα ταμεία αυτά είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα με τα συντακριτικά ταμεία, τα οποία παγκοσμίω ε, ε, διαχειρίζονται 35-3 δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για τριπλάσιο όγκο σε σχέση με τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Και βλέπετε στην πρωτοπινέκα από το Δεκέμβριο του 2015 ο συνολικός όγκος δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Τα κρατικά ταμεία και για το πετρέλαιο και για το αέριο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Παρά το γεγονό ότι υπήρξε τέτοια πτώση μεγάλη στι τιμέ του πετρελαίου και του αερίου. Και αυτό επειδή οι χώρε είχαν χρησιμοποιήσει καταρχά πρώτα τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και πρώτα πούλησαν τα κρατικά ομόλογα που υπήρχαν εκεί και προσπάθησαν στο βαθμό του δυνατού να κρατήσουν τους πόρους τους στα κρατικά επιμετικά ταμεία και ο συνάδελφος του πρώτου ομιλητή που ήταν υπεύθυνο του Νορβηγικού Επιμετικού Ταμείου είπε πρόσφατα ότι ενδεχομένω να μην υποστηρίζονται από τα επιμετικά ταμεία οι τιμές ε, των προσιακών στοιχείων αλλά παράλληλα αυτά πιστεύω ότι θα, ξανα, ότι θα εξακολουθούν να διδραματίζουν αντικυκλικό ρόλο και να αντισταθμίζουν την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πρώτες φάσεις της κρίσης του 2008 και 2009 τα κρατικά επενδυτικά ταμεία συνέβαλαν με παράδοξο τρόπο στην σταθερότητα των διεθνών αγορών. Βοήθησαν στην ανακεφαλοποίηση, για παράδειγμα, κάποιων μεγάλων τραπεζών όταν υπήρξαν μεγάλες απώλειες. Και γενικότερα συχνά κράτησαν τις αγορές σε επίπεδα καλός, καλής λειτουργίας, αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία, ενώ αλλά τα μία υποχωρούσαν. Άρα, γενικά, παρά το γεγονός ότι υπήρξε δραματική συρρήκνωση των πετρελαγορών, για παράδειγμα, και ε, έχουμε φτάσει σε επίπεδα ελλείμματος, υπήρξε μεγάλη αποθεματικό από τις κεντρικές τράπεζες και δεν ε, σημειώθηκε συρρήκνωση των κρατικών επενδυτικών ταμείων που ναι μεν σταμάτησαν να αναπτύσσονται και να διοικώνονται αλλά δεν συρρήκνωθηκαν και όλα. Και έτσι ε, καλύπτεται το δημοσιονομικό κενό με αγοραπολισίες ε, που γίνονται σε εύστοχο και επικαιρές χρονικές στιγμές και μακροπρόθεσμα ακολουθούνται πιο επικερδείς στρατηγικές παρά το γεγονός ότι ε, δεν υπάρχει μεγάλη επιρροή πλέον των ταμείων αυτών. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για τις διάφορες πηγές κρατικών επενδυτικών ταμείων και σε ό,τι αφορά την ε, αύξηση του κεφαλαίου τους. Και εδώ αναφέρομαι στο δεύτερο πίνακα που βλέπετε στην παρουσίαση μου, ένα μικρό πίνακα, τον υπαριθμό 2, και είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουμε με τους τρέχοντες λογαριασμούς. Ένας από τους βασικούς λόγους που υπάρχουν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία είναι τα πλεονάσματα των λογαριασμών. Και εδώ βλέπουμε διάφορα κίνητρα, διάφορους λόγους. Καταρχάς υπάρχει ο λόγος και το κίνητρο της ε, υποκατάστασης του πλούτου. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ε, την ε, αντικατάσταση ενός ε, φυσικού πόρου, σε περίπτωση, για παράδειγμα, στην περίπτωση του πετρελαίου. όπου ένας φυσικός πόρος ε, ε, μετατρέπεται ουσιαστικά σε επενδυτικό ταμείο, σε επενδυτικό πόρο. Άρα υπάρχει λόγος για μια αναπτυσσόμενη αγορά να παραμένουν οι πόροι αυτοί στο έδαφος όταν μιλάμε για απλή κατανάλωση. Αλλά οι εγχώρισες επενδύσεις στον πόρο αυτό έχει νόημα γιατί δημιουργεί ε, συσσόρευση κεφαλικών περιουσιακών στοιχείων για να υπάρξει μακροπρόθεσμα θετική επίδραση και στήριξη της εγχώρης οικονομίας. Και αυτό ισχύει προφανώς και για τις μακροπρόθεσμες, τα μακροπρόθεσμα ε, συνταξιδοτικά ταμεία. Έχουμε και φυσικά την ε, υπερβολική κατανάλωση των πόρων ή την ε, υπερπενδυση στις, σε κάποιες δομές για, κοινωνικές, ε, για κοινωνικά αφελη Η χρήση των εισοδημάτων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε χώρια είτε παγκόσμια και η απόφαση να εξαχθούν ή να μην εξαχθούν οι φυσικοί πόροι και η χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών θα πρέπει να επηρεάζονται από το επίπεδο εισοδημάτων της χώρας. Μια πλούσια χώρα όπως η Νορβηγία προτιμά προφανώς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποταμιεύσεις γιατί ο κόσμος είναι ήδη αρκετά πλούσιος. Μια φτωχή χώρα μπορεί να προτιμήσει να χρησιμοποιήσει τους πόρους για άμεσες επενδύσεις με άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά προφανώς συνδέονται και σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους. Ένας δεύτερος ε, λόγος είναι το πλεονάσμα των τρέχοντων λογαριασμών. Εδώ λοιπόν μιλάμε για χώρες όπως η Κίνα, άλλες χώρες της Ασίας, αλλά και τη Γερμανία ενδεχομένω, την Ολλανδία, που έχουν πλεονάσματα σε σχέση με το ΑΕΠ τους. Αυτά τα πλεονάσματα λοιπόν είναι αρκετά ανθεκτικά, αυξάνονται και αντέχουν και στι συναλλαγματικέ συνταραχέ. Η, τρίτος, η τρίτη αιτία είναι η αντικυκλικότητα. Έχουμε λοιπόν κυκλικές μεταβλητές, μετα, ε, βολές στις εξαγωγές και έχουμε και κυκλικές μεταβολές στις ε, τιμές. Όταν υπάρχουν διάφορες πηγές, ε, αυτό είναι δύσκολο σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της σταθερότητας, γιατί είναι δύσκολο να ξέρει μια χώρα κατά πόσον είναι μετα... προσωρινές ή μη οι μεταβολές αυτές και οι ασταθείς αυτές μία τεταρτή αιτία. Είναι η αυστηρή αιτία της ε, αυτοασφάλισης. Επειδή λοιπόν οι κεφαλαίκες ροές είναι κύκλικες αρχικά και στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, πιστεύαμε ότι τα κριτήρια τα σχετικά είναι η ανατρεψιμότητα των κεφαλικών ε, ροών. Στον δεύτερο λοιπόν πίνακα, όπως σας είπα, υπάρχει μια σύνοψη των διαφόρων αιτιών που καθορίζουν τη φύση των ταμείων που θα πρέπει να χρησιμοποιείται και την ε, ε, σύσταση των επενδύσεων. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επενδύσεις οι οποίες είναι πιο ενδεδειγμένες όταν υπάρχει πλεόνασμα και όταν υπάρχει μακροπρόθεσμη επιθυμία μακροπρόθεσμης απόδοσης. Κάτι άλλο που είναι σχετικό είναι το θέμα της στρατηγικής ε, χώρισης ε, περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάλογα με την προέλευση των πλεονασμάτων, γιατί είναι πιο σημαντικό αυτό από την ρευστότητα. Είναι πιο σημαντικό κατά πόσο είναι μακροπρόθεσμα και πιο μόνιμα τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και ως εκ τούτου ενδεχομένω να υπάρχει πολύ πιο μακροπρόθεσμος ορίζοντας και μικρότερη ε, προτιμήση για τον κίνδυνο από, τη, από πλευράς των πλούσιων ατόμων. Και γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένω να είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Να είναι λιγότερο κερδοσκομικά, αν θέλετε, λιγότερο βραχυπρόθεσμα σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν α, οι προηγούμενοι μιλητέ σε σχέση με τον α, ιδιωτικό, τον ιδιώτη επενδυτή. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και να μην χρησιμοποιούνται ε, τάχα άλλα, άλλη στόχοι πλασματικοί. Επίσης, λοιπόν, έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο είναι ευκταίο για όλα τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Τέλος, να αναφερθώ στο πόσο αυτά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να διοικητευτούν και να αποτελέσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Όπω σα είπα, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία είναι ιδανική φορήση για επενδύσει σε υποδομέ, ιδιαίτερα σε πράσινε υποδομέ σε καινοτομικέ υποδομέ. Μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ, το οποίο συνεπάγεται ότι οι επενδύσει στην, ε, στις υποδομές ε, είναι ενδεδειγμένες και εξασφαλίζει απόδοση, συντελεστή απόδοση που είναι αναλογικός με το τμήμα, με την δέσμευση που αναλαμβάνεται. Η μακροπρόθεσμη φύση των ε, ταμείων αυτών είναι ενδεδειγμένη για μακροπρόθεσμες τέτοιες επενδύσεις σε υποδομές. και έτσι υπάρχει λιγότερη έκθεση σε λιγότερο ρευστέ κατηγορίε ταμείων. Αυτό διευκολύνει την χρήση των κρατικών επενδυτικών ταμείων και υπάρχουν ήδη μεγάλοι επενδυτέ σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, για παράδειγμα, αλλά στο βαθμό που υπάρχει μεγαλύτερη ε, ζήτηση για επένδυση από την ΕΤΕΠ, από το ΕΦΣΙ, στην πλαίσια του σχεδίου Juncker, φαίνεται ότι τα κρατικά μέτρα τα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και να συμβάλλουν για να υπάρξει μεγαλύτερα προσιακά στοιχεία, μεγαλύτερε πόρη. Τρία θέματα κλείνοντα. Ενδιαφέροντα. Καταρχά, κατά πόσον θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικοί μηχανισμοί για να προσελκυθούν ε, κρατικά επενδυτικά ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα. Ο ρόλο των Κινέζων ε, επενδυτών στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Ενδεχομένω η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων να διαφερθεί να κάνει επενδύσει στην Ευρώπη. Κατά δεύτερον, οι εθνικές ε, τράπεζες ε, προώθηση, ανάπτυξης, Προφανώς ε, θέλουμε να παίξουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Σταγικών Επενδύσεων και σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχουμε από διάφορες τέτοιες τράπεζες στην Ευρώπη. Τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν λοιπόν αυτές οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες Ανάπτυξης και τέλος πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σαφώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια χρήσιμη πηγή για περαιτέρω χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Υπάρχουν τώρα συγκεκριμένοι μηχανισμοί που πρέπει να αναπτυχθούν για να γίνει αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα και επιπλέον αυτό πιστεύω ότι δεν συζητιέται επαρκώ. Διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν μεγάλα πλεονάσματα. 10-15%, συγγνώμη, 9-10% του ΑΕΠ του. Πώ θα μπορούσαν λοιπόν αυτέ οι μακροπρόθεσμε αποταμιεύσει να διοικητευτούν σε παραγωγικέ επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στι χώρε του, είτε σε άλλε χώρε, ιδιαίτερα μέσω μηχανισμών όπω το σχέδιο Juncker. Η Γερμανία, για παράδειγμα, τα γερμανικά και ολλανδικά συνταξιδοτικά ταμεία που έχουν μεγάλη κλίμακα θα μπορούσαν να επενδύσουν σε άλλε χώρε και ποιοι θα είναι οι καλύτεροι μηχανισμοί και τα καλύτερα κίνητρα που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Θα ήθελα να κάνω μια συντομή αναφορά και στο εξή. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, θεσμικά όργανα όπω η ΕΤΕΠ να δίνουν εγγύηση στον ιδιωτικό τομέα, όπω και προηγουμένω. Είναι σημαντικό, εξίσου σημαντικό, να αποφύγουμε τις διαρκείς και υπερβολικές εκθέσεις στην ιδιωτική αγορά σε περίπτωση δυσμενών συνθήκων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές. Και ερχόμαστε σε ερωτήσεις και απαντήσεις με τους ευρωβουλευτές. Δύο λεπτά για την κάθε ερώτηση. Πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας, παρακαλώ. Και μετά, σε τρία λεπτά, οι ομιλητές θα μπορέσουν να απαντήσουν. μέρος του Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εσάς ε, για το γεγονός ότι βρίσκεται μαζί μας σήμερα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, λοιπόν, Έχουμε διάφορα παραδείγματα επιτυχών κρατικών επενδυτικών ταμείων. Έχουμε εδώ εκπροσώπους της Νορβηγίας, για παράδειγμα, οι όροι λοιπόν εκεί είναι πολύ συγκεκριμένοι και ιδιαίτερη για κάθε διαφορετικό κρατικό επενδυτικό ταμείο και πιστεύω ότι η επιτυχία στον τομέα αυτό δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από χώρα σε χώρα και να μεταφερθεί από χώρα σε χώρα. Μία ερώτηση να κάνω προς τον κύριο Βάμπρακ, τον Υφυπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας. Μπορείτε κύριε Υπουργέ να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα να μας δώσετε μια επισκόπηση των όρων που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητοι για να υπάρχουν μακροπρόθεσμα επιτυχή κρατικά επενδυτικά ταμεία και να μπορούν και να τα συστήσουμε, να τα δημιουργήσουμε, αλλά και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε σε βάθος χρόνου. Και επίσης να ρωτιέμαι κατά πόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω καλύτερους, πιο ευνοϊκούς όρους για τη δημιουργία τέτοιων κρατικών επενδυτικών ταμείων. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει τώρα προς όλους τους πανελίστες. Τι γίνεται όταν υπάρχει ένταση μεταξύ των πολιτικών στόχων που τίθενται για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και φυσικά των οικονομικών ζητημάτων από την άλλη. Πάντα θα υπάρχει κάποια στιγμή τέτοια ένταση, κάποια σύγκρουση αν δεν υπάρχει ενδεχομένω η απόδοση που αναμένεται. Τι πιστεύετε για το θέμα αυτό. Please. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Έχουμε κάποια εμπειρία βέβαια από το δικό μας το επενδυτικό ταμείο πρώτα απ' όλα και νομίζω ότι κάποια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία είναι πρώτα απ' όλα να έχει κανείς σαφή στόχο για το τι θέλει από το επενδυτικό του ταμείο. Είναι καθαρά οικονομικός ο στόχος Είναι δύσκολο να έχει κανείς ένα επενδυτικό ταμείο με διαφορετικούς στόχους, με πολλούς και διαφορετικούς στόχους. Δεύτερον, χρειάζεται διαφάνεια. Είναι ζωτική σημασία για ένα επενδυτικό ταμείο. Η διαφάνεια απέναντι σε μια ανοιχτή κοινωνία, όπως έχουμε στις ευρωπαϊκές χώρες. Με πλήρη αναφορά όλων όσων συμβαίνουν στο Ταμείο. Έτσι μόνο υπάρχει εμπιστοσύνη από τους ιδιοκτήτες. Και τρίτον, να υπάρχει σαφής διάκριση ρόλων ανάμεσα στο Υπουργείο που εκπροσωπώ εγώ εδώ, που δίνει τις κατευθυντήριες ε, γραμμές και μετά από την άλλη να υπάρχει η διαχείριση, ο διαχειριστικός ρόλος που πρέπει να είναι διακριτός. Ευχαριστούμε. Η επόμενη απάντηση. Ναι, για να απαντήσω και εγώ για το θέμα αυτό της συμφωλίωσης του πολιτικού συμφέροντος με την απόδοση. Αν το επενδυτικό κρατικό ταμείο επενδύει κάπου συγκεκριμένα, αν είναι μακροχρόνια η φύση τους, τότε μπορεί να περιμένει να έχει παρετέρω υπόδοση και να επενδύσει από αυτά τα οποία θα έχει κερδίσει. Τα περισσότερα τέτοια επενδυτικά ταμεία επενδύουν σε equities ή σε ομόλογα. Αυτά που επενδύουν σε υποδομές ή ε, σε οικοδομικές δραστηριότητες, φυσικά ισχύει κάτι διαφορετικό. Και εσείς. Ναι, νομίζω και εγώ όπως όλες οι ερωτήσεις για το θέμα είναι δύσκολες εδώ. Μπορεί κανείς να κάνει τη διάκριση πολιτικά, αν το ερμηνεύσουμε στενά, μπορούμε να το δούμε σε μια χώρα, σε μια ομάδα χωρών. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και καλοί πολιτικοί λόγοι όπως η Νορβηγία, η οποία φροντίζει για τη βιωσιμότητα, για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους χρήστες του Ταμείου. Συχνά υπάρχει μεγάλη επικάλυψη των πολιτικών στόχων και των εμπορικών. Όταν δεν υπάρχει επικάλυψη, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κρατική χρηματοδότηση, αν ας πούμε ένα σχέδιο πράσινο είναι καλό και μπορεί να αποδώσει, μπορεί κάλλιστα να στοχεύσει σε αυτό και να επενδύσει εκεί ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, γιατί στο κάτω-κάτω είναι κοινωνικά αποδεκτό, εφόσον βέβαια υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Γίνεται δηλαδή και έτσι μπορούμε να ισορροπήσουμε τους δύο αυτούς στόχους, τον πολιτικό και τον οικονομικό. Φυσικά πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση στο επενδυτικό ταμείο. Αλλά πρέπει να είμαστε και αυστηροί από την άλλη μεριά με τους ιδιωτικούς επενδυτές που σωστά λένε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Δεν ζητάνε όμως το ίδιο από τα hedge funds. Εκεί μπορεί να μην έχουμε διαφάνεια. Οπότε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρέπει να κοιτάω και το ρολόι γιατί έχουμε και ψηφοφορία μετά. Λοιπόν, η υπερβάνος ε, Περέζη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τόσα μας είπατε για ένα θέμα που δεν εξετάζουμε πολύ συχνά εδώ στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας, το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο πρέπει να παρεύουμε με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στο πώς θα εξελιχθούν τα κρατικά αυτά επενδυτικά ταμεία. Στην αρχή της κρίσης είχαμε έναν πρώτο προβληματισμό και τώρα διαπιστώνουμε ότι λίγα πράγματα έχουν επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που εμένα ε, με ενδιαφέρει είναι το εξή. Μιλάμε για τα επενδυτικά ταμεία ω επενδυτέ, επειδή επενδύουν. Και ένα θέμα που δημιουργεί μεγάλη αίσθηση είναι όταν υπάρχει μια επενδυτική στρατηγική τέτοιου κρατικού επενδυτικού ταμείου, η οποία απειλεί την ε, κυριαρχία κατά κάποιο τρόπο και που επιτρέπει να κυριαρχήσουν τα συμφέροντα μιας χώρας. Δεν ξέρω είτε πρόκειται για διαδικασίες ιδιωτικοποίησης μεγάλων υποδομών κτλ. Όταν βρίσκονται στα χέρια επενδυτικών ταμείων δεν είναι πάντα φιλικά αυτά τα επενδυτικά ταμεία. Και στην Αμερικανική νομοθεσία υπάρχει μηχανισμός κατάλληλος που επαληθεύει τι γίνεται. Μήπως λοιπόν και η Ευρώπη θα έπρεπε να διαθέτει έναν αντίστοιχο μηχανισμό. Και από πλευράς διαχείρισης των πόρων, από τα ταμεία αυτά, τα ταμεία που επενδύουν στην Ευρώπη δεν θα έπρεπε να υποχρεθούν να συμπεριφερθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο ή η νομοθεσία που διαθέτουμε είναι παρκής. Η ερώτησή μου είναι και για τους τρεις αλλά υποθέτω ότι θα αποφασίσετε εσείς ποιος θέλει να απαντήσει στην ερώτησή μου. Πρόεδρος, ωραία, ποιος θα απαντήσει. Παρακαλώ. Αποφασίστε εσείς πριν αποφασίσω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Φαμράκ. Ναι, αυτά που ρωτάτε δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το Νορβηγικό Επενδυτικό Ταμείο. Γιατί εμείς έχουμε μικρά κομμάτια της κάθε εταιρεία. Και υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που λένε ότι καμία επένδυση σε equities δεν πρέπει να είναι πάνω από 10% της εταιρεία. Δηλαδή ποτέ δεν θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται. Αλλιώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για τα equities έχουμε αυτό τον περιορισμό. Τώρα, σε επενδύσεις στο νοικοδομικό τομέα, και εκεί έχουμε ρύθμιση. Και αν κάποιος θέλει να επενδύσει σε μη σαγμένες υποδομές, θα πρέπει να είναι πάνω από 10% το ποσοστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, μια κυρία Γκρίφιτ Τζόνς. Και πάλι εξαίρετη ερώτησή σας. Θα μπορούσε κανείς να βάλει προϋποθέσεις. Εάν ιδιωτικοποιηθεί μια εταιρεία, για παράδειγμα, πρώτον υπάρχει η τιμή η οποία θα πρέπει να ανακριβείς. Δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει η επένδυση αυτή να συνδυαστεί με νέες επενδύσεις και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι απλώς ότι προσπαθεί κανείς να αγοράσει φτηνό κεφάλαιο. Όχι. Αυτό βοηθάει τις επενδυτικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται νομοθεσία γι' αυτό ή κίνητρα, πάντως θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε νέες επενδύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και ο Κίντο. Ναι, πολύ σύντομα. Πράγματι είναι βασική ερώτηση αυτή και έχει να κάνει με το θέμα της διαφάνειας χαρακτηριστικά. Πρέπει κανείς να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε περιουσιακό στοιχείο εμπορεύσιμο και μη εμπορεύσιμο. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί κανείς νομοθετικά να καθορίσει ένα το ποσό επενδύσεων σε ένα μέσο. Για τις equities, για παράδειγμα, ποσοστό ιδιοκτησία, αλλά και σε άλλες συναλλαγές θα μπορούσε κανείς να περιορίσει το ποσό με ένα ποσοστό απέναντι σε ομόλογα κλπ. Στην άλλη περίπτωση, τα μη εμπορεύσιμα είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Εδώ το ζήτημα κλειδί είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τα μέσα και ποιες είναι οι κλείδες ασφαλείας από τις οποίες απορρέει η ανεξαρτησία τελικά των ε, περιουσιακών αυτών στοιχείων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θέλετε το λόγο από το ECR, Λούκη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Ένα τέτοιο κρατικό ταμείο χρησιμοποιεί κρατικές, ε, κρατικές δαπάνες, τα οποία και δαπανούνται για κάποιους σκοπούς. Η εναλλακτική χρήση των ε, κρατικών δημοσίων αυτών πόρων είναι να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα του κράτους, είτε είναι από φόρους, είτε είναι από πρώτες ύλους, να επιστραφούν στους πολίτες μέσω μείωσης των φόρων. Άρα ουσιαστικά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία θεωρώ ότι είναι μια υποχρεωτική ουσιαστικά συσσόρευση πλούτου που δεν είναι όμως ε, ε, δεδομένο ότι έχει πολιτική υποστήριξη. Πρόκειται για ένα αγαθό το οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, όποιος αποφασίσει να δημιουργήσει κρατικά μυθικά ταμεία και έτσι σημαντικοί πόροι επενδύονται στα πλαίσια των ταμείων. Αυτό, αυτό προφανώς ε, υποστηρίζεται από τον κόσμο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν υποθέσουμε και θεωρήσουμε ότι πρόκειται για οικοδόμηση για δημιουργία τέτοια ε, πλούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κρατικά τα ταμεία στην κεφαλαία αγορά και να, δο, να οριστούν ε, πιστοποιητικά προκειμένου να είναι δεδομένο ότι υποστηρίζονται από τον κόσμο γιατί ενδεχομένω κάποια τμήματα του κόσμου να θέλουν να έχουν πιο πολλέ τέτοιε επενδύσει και ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουν και δυτικού πόρου, αλλά ενδεχομένω και η απόδοση που θα έχει ένα τέτοιο ταμείο να είναι ελκυστική σε κάποιες ε, τέτοιου καιρού που είναι δύσκολο να έχουμε θετική απόδοση των ταμείων. Έχετε σκεφτεί λοιπόν να ανοίξετε και να συμπεριλάβατε και ιδιωτικά επαρκούς πόρου στα κρατικά επενδυτικά ταμεία ενδεχομένω και για την πραγματοποίηση αμφιλεγόμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να απαντήσει. Είμαι γενναία. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Λόγω χάρη Κινέζικη κυβέρνηση και άλλες Κάποια από τα περιουσιακά του στοιχεία δεν ξέρω αν από το θεματικό τους ή από τα SWF, έχουν ε, χρησιμοποιήσει τους πόρους για να δημιουργήσουν την ε, Ασιατική Τράπεζα Υποδομών. Κάτι ανάλογα έκανε και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τη δεκαετία του 50, που πήραν τους πόρους τους και χρησιμοποίησαν το κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το αυγάτισαν. Βεβαίως δανείστηκαν και από την αγορά κεφαλαίων. Ε, έτσι παίρνει κανείς μόχλευση από ε, τις αγορές κεφαλαίων, όπως με το ΕΦΣΙ και τη μόχλευση του 15%. Με άλλες τράπεζες λοιπόν, με συγχρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από ιδιώτες επενδυτές, έτσι γίνεται. Ε, και το βρίσκω καλό, διότι περνάει κανείς από δοκιμασμένα ιδρύματα και αρχές. Όμω, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα τα SWF ευθεία να δανείζονται. Διότι θα δημιουργήσουν ε, δυσκολίε ε, με τη ροή κεφαλαίων ή τις σχετικέ επενδύσεις και αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειε. Αυτό που είναι όμορφο στο, στα SWF είναι ότι είναι μακροπρόθεσμε οι επενδύσεις. Μπορεί κανεί να επενδύσει δηλαδή για το πολύ απότερο μέλλον. Ευχαριστούμε. Το δικό μας SWF βεβαίως ε, βασίζεται στις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου, από εκεί έχουμε πάρει τα εισοδήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα εισόδημα που δεν μπορεί να ανανεωθεί προς την κυβέρνηση. Η σύμβασή μας με τον πληθυσμό είναι ότι θα εξορίσουμε αυτού τους πόρους για ένα σύντομο διάστημα και θα υποφεληθούν περισσότερες γενιές πολιτών από αυτό το εισόδημα από όσους τώρα βρίσκονται εν ζωή. Από την σκοπιά λοιπόν του πληθυσμού ε, η σύμβασή μας, η συμφωνία μας βασίζεται ακριβώς σε αυτήν την λογική ότι οι δαπάνες γίνονται με σκοπό το απότερο μέλλον με μείωση των φόρων για μια-δυο γενιές, κάτι που θα επιτρέψει να υπάρξει ευημερία και ευμάρεια για πάνω από μια γενιά. Το SWF λοιπόν μετράει και στο ΕΠ μας, είναι ένα μεγάλο μέρος του. Τώρα βέβαια θεωρητικά μπορεί να προσθεθεί κεφάλαιο από την ιδιωτική αγορά στο Ταμείο. Και πάλι όμως δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από το στόχο του Ταμείου. Δηλαδή θέλουμε και να ε, μεγαλώσει το κεφάλαιο, αλλά και να προστατεύσουμε αυτά τα κεφάλαια για το μέλλον του νορβηγικού πληθυσμού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μονό από το ΕΝΕΦ e τώρα. Καλησπέρα στους προσκεκλημένους. Ευχαριστώ που ήρθατε. Η ερώτησή μου είναι, κύριε Υφυπουργέ, ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ των SWF και των κρατικών χρεών. Ξέρουμε πολλές φορές ότι οι δημόσιες πολιτικές καθορίζονται από αυτά τα ταμεία. Όμω μπορεί οι δραστηριότητε μια εταιρεία σε μια χώρα να έχουν πολύ μεγάλε συνέπειε. Το Ταμείο τη Μέση Ανατολή και τη Ασία είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο, αν ε, εξαιρέσουμε την Ορβηγία τη χώρα σα. Πιστεύετε ότι τα SWF είναι ένα παράδειγμα και μια απειλή, διότι παράδειγμα, όπω στη χώρα μα, είναι ότι ένα μέρος του εισοδήματο από τα πετρέλαια, από το πετρέλαιο και τις εκαγωγές που το χρησιμοποιούν για τα ορεκτά καύσιμα και λέτε ότι γίνονται επενδύσεις μακροπρόθεσμες. Αυτό μπορεί να αποσταθεροποιήσει την οικονομία. Μπορεί όμως να είναι και απειλή. Όταν οι ξένες επενδύσεις είναι μαζικές και μπορεί να ε, ε, θέσουν ένα αμφιβόλο την ανεξαρτησία ενός έθνου. Αυτό με το ΚΑΚ 40, το δίκτυο του χρηματιστηρίου της Γαλλίας, όπου υπάρχουν πολλές τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Αυτό λοιπόν ήθελα να ρωτήσω. Στις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις, η πολιτική ε, διάσταση, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει, ιδίω ε, στην αγορά αξιογράφων, και τι ορίζοντα προβλέπετε για τη συμμετοχή σε διάφορες εταιρείες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τη διαχείριση και αυτό σας οδηγεί να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη δίκη σε μιας επιχείρησης. Δηλαδή, μπορείτε να είστε ένας μέτοχος που ε, εξασκεί επιρροή. Επίσης, εξαιρείται από το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο κάποιες ε, ε, εταιρείε, όπως τις εταιρείε ορυκτών καυσίμων, τον άνθρακα, τα περινικά και των όπλων. Επίσης δεν δέχεστε δημόσια εταιρείες που αμείβουν ε, πολύ ψηλά ποσά τους εργοδότες τους, τα υψηλά στελέχη ή έχουν μεγάλες απώλειες στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν έχει κάποια σημασία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στην ερώτηση για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ναι, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του διαχειριστή των SWF της Norske Bank. Πρώτα απ' όλα έχουμε οικονομικό στόχο μεγιστοποίησης των οικονομικών μας επιστροφών με κάποια όρια για την έκθεση σε κίνδυνο η αξιολόγηση γίνεται από την Norske Bank, την κεντρική μας τράπεζα, σε ό,τι αφορά το ότι αποφέρουν τα ομόλογα λόγω χάρη και η τράπεζα είναι υπεύθυνη για το ποιες εταιρείε θεωρούνται καλέ ή όχι για επενδύσει. Έχουμε όμως και κάποια διοντολογία, κάποιες αρχέ διαδολογίες που μας κατευθύνουν. Δηλαδή τι μπορεί να διαχειριστεί και να αποφασίσει να επενδύσει, σε τι πρέπει να αποφασίσει να επενδύσει η Norske Bank. Είπατε τα πυρηνικά όπλα και ούτω καθεξής που ε, είναι κάτι που αφορά και τον νορβηγικό πληθυσμό. Δεν θέλουμε να ε, έχουμε εισοδήματα από την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής ή πυρηνικών όπλων. Αυτά αποκλείονται από το επενδυτικό μας περιβάλλον. Και εταιρείες με αντιδεοντολογική ε, συμπεριφορά και πρακτικές που έχει αποδειχθεί συν το χρόνο επίσης αποκλείονται. Υπάρχει κριτήριο αποκλεισμού τα οποία το επιβάλλει και το Υπουργείο. Είναι εταιρείε τι οποίε η τράπεζα δεν μπορεί να επενδύσει. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανεί άλλο το λόγο. Επόμενο για το ΕΛΚ ο κύριος Στόλογιαν. Σα ευχαριστώ. Έχω τρει ερωτήσει. Η πρώτη προ ε, τον εκπρόσωπο της ε, Νορβηγία για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Είπατε ότι η Κεντρική Τράπεζα η οποία διαχειρίζεται τα κρατικά επενδυτικά ταμεία έχει μία εντολή από τον Υπουργό Οικονομικών. Αν έχει λοιπόν εντολή από τον Υπουργό Οικονομικών, πρέπει να λογοδοτεί και στον ε, Υπουργό Οικονομικών. Είναι λίγο περίεργο αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τη σχέση μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και ε, του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι υποτίθεται ανεξάρτητα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ειδική, ειδικές γνώσεις για τις κεντρικές τράπεζες. Υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό τμήμα με τέτοιου είδους εμπειρογνωμοσύνη, φαντάζομαι. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο... Πώς τον Κύριο Ματσίζιο, τον Γκουίντο Ματσίζιο. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία. Έχουμε μια μεγάλη ιστορία για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται, να δεν χάνουν διαχείρισης οι κρατικές ε, εταιρείε. Έχουμε οργανισμούς για τη διαχείριση των ε, εταιρείων αυτών με εντολές κτλ. για τη διαχείριση αυτών. Τώρα έχουμε και μια νέα ιδέα από τα κρατικά αυτά επενδυτικά ταμεία. Υπάρχει μια ιδέα των κυβερνήσεων προκειμένου τα κρατικά επενδυτικά ταμεία τα οποία αφενός θα διαχειριστούν και την κρατηματική συμμετοχή σε κρατικές επιχειρήσεις και ένα νέο χαρακτηριστικό να επενδύει. Δυστυχώς. Το ερώτημά μου είναι γιατί είναι καλύτερο να πάρουμε πόρους που δεν σχετίζονται με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, όπως είναι στην Νορβηγία. Έχετε υψηλέ τιμές για το πετρέλαιο και αποφασίσατε να συστήσετε ένα τέτοιο κρατικό επενδυτικό ταμείο. Αλλά γιατί να λάβουμε απόδοση από όλε, να πάρουμε πόρου από όλα τις κρατικές εταιρείες και να επενδυθούν. Γιατί να είναι καλύτερο αυτό σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, σε ό,τι αφορά άλλα στοιχεία και προβλήματα που μας απασχολούν. Γιατί να μην μείνουν οι πόροι αυτοί στον κρατικό προϋπολογισμό και να λεφθούν οι αποφάσεις ε, για τις κρατικές δαπάνες μέσω του κοινοβουλευτικού, της κοινοβουλευτικής οδού. Ξέρετε επίσης ότι μπορεί να υπάρχει έλλειμμα τρέχων λογαριασμών, αλλά το ερώτημα που έχω να κάνουμε είναι σε ποια κατάσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διεθνείς πόρους που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των εθνικών τραπεζών για να χρηματοδοτηθούν τέτοια κρατικά την ταμεία. Πολλές ερωτήσεις, παρακαλώ. Οι απαντήσεις ήταν σύντομες όμως. Να προσπαθήσω να διευκρινίσω ποια είναι η σχέση μας με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε δύο διαφορετικές ε, σχέσεις πέρα από την νομισματική πολιτική η Κεντρική Τράπεζα είναι εντελώ ανεξάρτητη από την από την Υπουργή Οικονομικών. Στον άλλο του ρόλο ως διαχειριστής των ταμείων, η Κεντρική Τράπεζα διαχειρίζεται τέτοια ταμεία για ιστορικούς κυρίως λόγους. Θεωρούμε ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι ο πιο ενδεδειγμένος διαχειριστής τέτοιων ταμείων. Και στη σχέση αυτή η διαχείριση των ε, ταμείων ανατίθεται σε ιδιαίτερο τμήμα α, της Κεντρικής Τράπεζας, ένα τμήμα που έχει μόνο ένα πελάτη, τον Υπουργό Οικονομικών. Και η σχέση αυτή λοιπόν ε, διαχειρίζεται από το τμήμα αυτό. Που δίδεται λοιπόν από την Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω το διαδικαστικό κομμάτι, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας. Αν θέλετε να δείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κρατικών επενδυτικών ταμείων, των θεσμών που τη διαχειρίζονται τέτοια ταμεία και του κύκλου του προπολογισμού, θα έλεγα ότι η βασική διαφορά έγκυται στο εξή. Η κατάρτιση του προπολογισμού υπόκειται σε ένα πολιτικό κύκλο, αν θέλετε. Αν θέλετε να υπάρχει ανεξαρτησία από τους πολιτικούς φορείς, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια διαρκής ε, και μακροπρόθεσμη συμφωνία και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, στην περίπτωση αυτή λοιπόν δημιουργείται, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δηλαδή, μία ανεξάρτητη αρχή. Αυτή η ανεξαρτησία έγκυται στα κριτήρια διαφάνειας, με σαφή λογοδοσία, με σωστή μέτρηση των αποτελεσμάτων και μετά μπορεί να υπάρχει διαχείριση όπως Νορβηγία για παράδειγμα από το Υπουργείο που θέτει κάποιες βασικές αρχές, αλλά μετά θα πρέπει να γίνει ανάθεση της διαχείρισης για να υπάρχει επιρροή στη διαχείριση των επενδύσεων. Να μην υπάρχει επιρροή δηλαδή των αποφάσεων που λαμβάνεται με ενδεχόμενη συγκρίση συμφερόντων από πλευρά των πολιτικών φορέων. Πρόκειται λοιπόν για μια. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, Πρόεδρε. Περιμένουμε και την τρίτη απάντηση, λέει ο Πρόεδρο. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, να είμαι σύντομη. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των τρέχων λογαριασμών και των κεφαλαιακών λογαριασμών. Αν στους τρέχοντες λογαριασμούς υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα, όπως για παράδειγμα έχει η Κίνα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση αυτή έχει νόημα να επενδεθούν τα στοιχεία αυτά. Αν υπάρχει ένα πλεόνασμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι προσωρινό και αυτό φυσικά είναι πιο δύσκολο στην πράξη να εκτιμηθεί, τότε θα έχει νόημα να διατηρηθούν σε αποθεματικό κάποιοι από αυτού τους πόρους. Και για να χρηματοδοτηθούν οι μελλοντικέ εισαγωγέ, τουλάχιστον τρει μήνε εισαγωγών, αυτό είναι ο στάνταρ κανόνα, αλλά και σε περίπτωση που οι κεφαλαϊκέ επιρροέ ε, αντιστραφούν. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια προσωρινή, βράχη πρόθεσμη μεταβολή. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να υπάρχουν τα πραγματικά αυτά. Και τέλος, και οι πολίτε ενδεχομένω να προκαλέσουν κεφαλαί... Ε, μάλλον εκρόγει των κεφαλαίων, των αν υπάρχουν ε, σχετικοί όροι και συνθήκες. Αν υπάρχει όμως μακροπρόθεσμα πλεόνασμα, όπως στη Γερμανία, στην Κίνα, καλά παραδείγματα και αυτά, έχει νόημα να μπουν τα πλεονάσματα αυτά σε κρατικά επενδυτικά ταμεία, σε εργαλεία και να αξιοποιηθούν είτε για επενδύσεις ε, στο εξωτερικό είτε για επενδύσεις χώρια για την διαφοροποίηση της οικονομίας προκειμένου να καταστεί λιγότερο εξαρτημένη. Ευχαριστώ πολύ. Από την ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Τάγκ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω προς τον ε, Υφυπουργό καταρχάς. Να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχάς ε, προωθεί ιδιαίτερα την ιδέα των, ε, της υπεύθυνη επένδυσης μέσω των κριτηρίων ESG, ιδιαίτερως. Στην οδηγία για τα στακριτικά ταμεία, για παράδειγμα, τα οποία εφαρμόζουν θελούσια σε κάποιες περιπτώσεις τις αρχές αυτές υποχρέωση λογοδοσία σύμφωνα με το δίκαιο. Τα νορβηγικά κρατικά βέβαια πώς συνδέονται με τα κριτήρια IC του ΟΙΕ και περιλαμβάνεται επίσης γιατί αυτό ασφαλώς μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνδέεται με το θέμα λοιπόν της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής. Την ημέρα που δημοσιεύθηκαν τα έγγραφα Πάναμα σε παγκόσμιο επίπεδο τα κρατικά παιδικά ταμεία έχασαν ε, σημαντικό τμήμα της αξίας τους λόγω των επενδύσεων σε εταιρείε που ήταν εμπλεκόμενες στα Panama Papers. Πείτε μας λοιπόν ε, πώς ε, υπάρχει επιρροή και στα νορβηγικά ταμεία προς την καθηγήτρια Griffin τώρα. σε ό,τι αφορά και την επιρροή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είπατε ότι θα μπορούσε η Γερμανία και η Ολλανδία να μειώσουν το πλεόνασμά τους εάν υπήρξε τέτοια επένδυση στα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία. Αυτή είναι η πιο σόφρον λύση. Μήπως υπάρχουν και πιο ανταδειγμένες ε, λύσεις. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την απάντησή σας. Uh, Ευχαριστώ. Η Νορβηγία επιθυμεί την διαφάνεια αυτή και επίσης κάποια ταμεία διαφόρων ειδών στρέφονται προς αυτές τις λύσεις και προς εμάς για να αντιγράψουν τα κριτήριά μας υπευθυνότητα. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, πρόκειται για μακροχρόνιες επενδύσεις και είναι σημαντικό για μακροχρόνιες επίσης αποδόσεις να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και κοινωνικά υπεύθυνοι. Επίσης όμως να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα και το θέμα της φορολογίας. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτησή σας. Υποστηρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν ε, τους φόρους τους στις χώρες υποδοχής Um, Νομίζω και εγώ ότι η ερώτησή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πάντα το έγραφα και τώρα με τον καθηγητή Στίγκλιτς ετοιμάζουμε ένα βιβλίο όπου λέμε ότι η πρώτη απάντηση είναι να μειώσουμε το υπερβολικό πλεόνασμα στους τρέχοντες λογαριασμούς σε χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία, κάτι το οποίο επηρεάζει όχι μόνο την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το πλεόνασμα αυτό για παράδειγμα σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο στη Γερμανία από ότι στην Κίνα και υπάρχει αποπλοθεριστικό αποτέλεσμα και επιπτώσεις. Για παράδειγμα, επενδύοντας περισσότερο για τη Γερμανία, παρόλο που οικονομικά ήταν τόσο αποτελεσματική, έχει πολύ χαμηλές επενδύσεις. Από την άλλη χρειάζεται και υποδομές, οπότε και αύξηση των μισθών επίσης. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει περισσότερες επενδύσεις. Αν αυξάνονταν οι μισθοί στη Γερμανία, η Γερμανία από τη δικιά τους την πλευρά θα μπορούσαν να πάνε περισσότερο διακοπές στην Ελλάδα, στην Ιταλία και θα μπορούσαν και να περάσουν όμορφα, αλλά και συγχρόνως αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό για την ελληνική και την ιταλική οικονομία. Οπότε είναι αυτό που ονομάζουν οι οικονομολόγοι μια κατάσταση win-win, από την οποία και δύο πλευρές έχουν να κερδίσουν. Βέβαια, το πρόβλημα θα ήταν ότι παρόλα αυτά θα παρέμενε υψηλό πλεόνασμα. Και το ενδιαφέρον ζήτημα εδώ είναι να γίνουν εμπορικές επενδύσεις και έχει κάνει κάποιες μεταφορές σε διαφορετικά ταμεία και τα λοιπά η Γερμανία, αλλά επενδυτικές, ε, μάλλον εμπορικές επενδύσεις θα έπρεπε να αποτελεί την προτεραιότητα στις περιπτώσεις αυτές και να γινόντουσαν αυτές οι εμπορικές επενδύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη ε, όπου θα κέρδιζε και εκείνη και όλοι. Γιάκο Φαν Βέιτσιγκερ έχει τώρα το λόγο. Δύο ερωτήσει έχω εγώ μετά από την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα. Η πρώτη μου έχει να κάνει με τον ρόλο που έχουν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία στην τροποποίηση του κρατικού δανεισμού προκειμένου αυτός να γίνει κρατικές επενδύσεις. Με μεγάλη διαφοροποίηση βέβαια, γιατί είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η Νορβηγία, ενώ έχει ένα τέτοιο ταμείο που είναι 2,5 φορές του ΕΠ έχει ένα χρέος της τάξης του 30%. Η ερμηνεία που θα μπορούσε κάποιος ε, να δώσει είναι ότι αντί να ξεπληρώσει το χρέος επενδύει ε, αλλού. Να έχει μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο και χαμηλότερη εξυπηρέτηση χρέους. Οπότε ρωτάω, οι ευρωπαϊκές χώρες όπου το κόστος επενδύσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό, δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, να πούνε δηλαδή ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ όρεξη για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, είτε ομόλογα, είτε εξορτία με υψηλές τιμές και τα χρήματα αυτά να τα πάρουν και να τα επενδύσουν όπως ε, κάνει και η Νορβηγία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη. Θα ήταν καλή ιδέα να επιτρέψουμε στους πολίτες οι οποίοι δυσκολεύονται στον ιδιωτικό τομέα να βρούνε τρόπους να επενδύσουν μακροπρόθεσμα με χαμηλό κόστος συναλλαγών, θα ήταν καλή να τους επιτρέψουμε να επενδύσουν στα κρατικά επενδυτικά ταμεία τα οποία εμπιστεύονται υποδομές ή άλλο και το ρωτάω βέβαια και στον Νορβηγό Υπουργό και σε οποιοδήποτε άλλο θα ήθελε να μου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι έχει νόημα για τις περισσότερες χώρες να έχουν ένα κάποιο επίπεδο χρέους για, οικονομικά, για οικονομικούς τεχνικά λόγους, για να έχουν ας πούμε μια αγορά για τα κρατικά ομόλογα. Αν δεν έχετε ομόλογα, δάνεια δεν έχετε αγορά, δεν έχετε τιμή αγοράς για τα ομόλογα στο νόμισμά σας. Έπειτα, για να επιτρέψουμε σε άλλες χώρες ή σε άλλους επενδυτές γενικά μιλώντας να επενδύσουν και αυτοί σε κρατικά επενδυτικά ταμεία. Εμείς δεν το βλέπουμε για το συνταξιδοτικό νορβηγικό ταμείο, αλλά άλλα ταμεία θα μπορούσαν να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Άλλος, κανείς, να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Το δεύτερο σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενθαρρύνουμε πολίτες να επενδύσουν μαζί με κρατικά επενδυτικά ταμεία. Εφόσον βέβαια μπορούν να αγοράσουν ομόλογα οι πολίτες. Δεν έχουν μεγάλες αποδόσεις, αλλά ε, αποφέρουν πολλά Οπότε μπορεί να είναι μια καλή επένδυση. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα το διευκόλυνε αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα ειδικό μηχανισμός όπως έχουν οι Άπωνες με ειδικού αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους και ομιλητές μας ο χρόνος όμως περνάει δυστυχώς. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι και σας και όλους τους συναδέρφους που παρευρέθηκαν. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον Πρόεδρό μας. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ Μάρκους. Πρώτα απ' όλα κάποιες ανακοινώσεις. Η πρώτη είναι μια πολύ θλιβερή ανακοίνωση. Έμαθα ότι χθε το απόγευμα, δυστυχώ, χάσαμε τον Κάντο Μπερέν, πολιτικό σύμβουλο της ομάδας Άλτε, εκ μέρους της Επιτροπής μας. Θα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας και την συμπόνια μας, την οικογένεια, τους φίλους και του συναδέλφους του. Κόρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Αυτού του είδους την ομιλία δεν θα θέλει ποτέ κανείς να έχει το καθήκον να την εκφωνήσει, αλλά θα θέλει να, παραθέσει, να παραθέσω τα λόγια του αρχηγού μας, τον κύριο Περχόφστα, το οποίο είπε ότι θα θυμάται πάντοτε τον Κόχο ως έναν αξιόλογο επαγγελματία, αφοσιωμένο στη δουλειά μας και πάντοτε ε, ενημερωμένο, γνωρίζοντας απολύτως τι συμβαίνει και ε, διεξοδικό στις λεπτομέρειες. Ε, δεκριτική, αλλά με αυτοπεποίθηση και όσο την γνωρίζαμε καλύτερα, θερμή στις προσωπικές της σχέσεις. Ε, έτυχαν σεβασμό από τους συναδέλφους της, συναδέλφους της είχε ψηλότατα προσόντα και ήταν μια επικοδηματική συνάδελφος. Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε την αγκάρδια συμπόνια μας προς την οικογένεια και τους συναδέλφους της και όλους εδώ που εργάστηκαν κοντά της. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να τηρήσουμε ένα λεπτό συγγύηση. Και τώρα συστάσεις και αποφάσεις των συντονιστών 11 Απριλίου. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ετοιμάσουν εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, για τον κανονισμό των ε, οικονομικών σχέσεων, την επίβλεψη και την βιώσιμα, τα βιώσιμα δημοσιονομικά, εκθέσεις λεύκανση παράνομων προσόδων, πράσινη, γνωμοδότηση 53 συν εντολές δίμευσης ΕΛΚ, συμφωνήσαμε επί της πρότασης για, για το διαχωρισμό, το fast tracking, ενώ οι συντονιστές αποφάσισαν να μην ε, προχωρήσουμε σε fast tracking για το κεκτημένο θα την δούμε ξανά αυτή την απόφαση αργότερα μάλλον για τα ΕΖΑ θα υπάρξει διάλογο με την κυρία Ροζιά, αυτό αποφάσισαν οι συντονιστέ. Για τα μέτρα επίπεδου 2, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ξεκινήσει η διαδικασία για αντίρρηση. για την πρόταση της 20ης Μαρτίου και τον κατάλογο των χωρών με ανεπάρκειες στα καθεστώτα EML ΕΡΕΦ ναι, δημόσιες αποφασίστηκε το πακέτο για τις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις CRD, RAF ε, και όλα τα σχετικά να διοργανωθεί σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη ενημέρωση για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις είχαμε τον πρώτο τρίλογο για την ε, securization την ομολογοποίηση τον Απρίλιο την τιτλοποίηση τον Απρίλιο και με εντολή βάσει του άρθρου 272 ή να υπάρξει εντολή για τη διαπραγμάτευση για την τιτλοποίηση και με το άρθρο 56K να υπάρξει ενδεχόμενος μεταρρύθμιση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να ζητήσουμε νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή αντί για κατεξοδότηση πράξη δύο εντολέ για το τεχνικό επίπεδο και την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 591, λαμβάνοντα υπόψη τι ανησυχίε του Συμβουλίου και του ΕΛΚ. Και μετά από τριετή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση μαζί με την νομοθετική πρόταση όπω ε, δει. Για τον κανονισμό SDS, οι συνομοθέτε ενέκριναν κάποιε τεχνικέ πρόοδου και τα κριτήρια ESG να συμπεριληφθούν στις προϋποθέσεις αποκάλυψης στοιχείων με περισσότερο πρακτικό τρόπο, όπως ζητήθηκε. Στο τεχνικό επίπεδο το άρθρο 28 αποφασίστηκε και αυτό να εκχωρηθεί. Και για τον κίνδυνο της κατοχής στοιχείων και των μικροοικονομικών απειλών αποφασίσαμε να ε, αξιολογήσουμε το επίπεδο κινδύνου και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί το non-paper για τη σχετική αγορά και την μικροπροληπτική πρόταση καθώς και την μακροπροληπτική. Το έγγραφο της Επιτροπής για την Εποπτεία για να διευκολυνθεί η ερμηνεία των κριτηρίων από την ΕΣΜΑ, ενώ θα ζητηθεί να υπάρξει μια κοινή επιτροπή ΕΣΜΑ-ΕΖΑ για να διευκολυνθούν όλα αυτά, θα προχωρήσει. Και για το άρθρο 17 και τις κυρώσεις, το θίξαμε αλλά δεν επετέχθη συμφωνία. Οι συνομοθέτες συζήτησαν το έγγραφο της Επιτροπής για τις απαιτήσεις διαφάνειας Θεωρήθηκε αποδεκτό τρόπο να ευθυγραμμιστούν οι προποθέσει που επιβαλλονται στου ε, κατόχου τυπλοποίηση. και οι ιδιωτικοί φορείς να ε, εξαιρεθούν από αυτό, χωρίς να δημιουργηθούν να Και τα εναποθετήρια αυτής της τιτλοποίησης να ε, ρυθμιστούν σωστά. Με συγχωρείτε για την τόσο μακροσκελή ενημέρωση, αλλά ήταν ε, απαραίτητο να σας δώσω τις λεπτομέρειες, γιατί υπήρξε διαφάνεια στην πρόοδο των θεμάτων και ε, προχωρήσαμε σε αυτόν τον τόσο σημαντικό φάκελο. Τι ωραία να προχωρήσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία μας. Ελπίζω να έχετε ετοιμάσει τις κάρτες σας για να κάνουμε τον έλεγχο. Εψήφισαν άπαντες. Ωραία. Να ψηφίσουμε όπω ξέρετε. Κόρα Φανίβενχόιζεν. Έκθεση για το FinTech. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ή ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, 185 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Κάποιοι καθυστέρησαν να σκόσουν τα χέρια του ήταν υπέρ. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Π υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται ψηφορία πέρας Απορρίπτεται. Συμβαστική Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 261. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΜΚΟ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΜΚΟ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I. Ένα, με συγχωρείτε, ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 45 υπέρ 6 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Επόμενη συνεδρίαση, Τετάρτη 3 Μαΐου, 9 με 12.30, 3 με 6.30. Η συνεδρίασή μας λίγη.